μπορούμε να εγκρίνουμε αυτή την εντολή. Οι ελληνικές αρχές μου ζήτησαν άρση της ε, ασυλίας του κυρίου Μανώλη Κεφαλογιάννη για να εκινήσουν μια διαδικασία ενώπιον της δικαιοσύνης.